Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Άρχεται η συνεδρίαση. Καθίσατε όλοι φαντάζομαι και βάλατε και τα ακουστικά σας. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι το υπαρίθμημα 12. Πριν όμως αρχίσουμε, θα ήθελα να σας πω ότι όχι το επόμενο θέμα, αλλά το 14 μετατίθεται. Να σας πω και για πότε. Μετά το 6, το οποίο 6 το είχαμε μεταθέσει χθες. Αλλά πάντα για σήμερα το πρωί είναι και το 6 και το 14 διότι ο κύριος Ντόιτς ε, είναι σε άλλη επιτροπή, απασχολημένος. Και τώρα ακολουθεί πάμε το 12. Ισόρροπη λέει εκπροσώψη των φίλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών. bitte, Frau... Παρακαλώ την κυρία Κορνέλισεν να λάβει το λόγο. Μαράια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τι να σας πω. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Έχουμε συζητήσει με πολλούς για αυτό το θέμα. Λίγα είναι τα θέματα που ξεσηκώνουν τόσα πάθη. Έχει γίνει μια πρώτη συζήτηση στην ε, ε, αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, στη Γιούρη και τη ΦΑΜ. Είναι δύο επιτροπές, ε, παρακαλώ. Έχει γίνει μεγάλος λόγος για το πώς ε, μπορεί να βελτιωθεί αυτή η πρόταση. Προσπαθώ και εγώ με τη σειρά μου να κάνω μερικές ε, βελτιώσεις και με περίεργη να ακούσω τι θα μου πείτε σχετικά. Τι κάναμε, κάτι μικρό, αλλάξαμε τον τίτλο, αλλά και κάποιους παραγράφους για να πούμε ότι καλύπτει και τις εκτελεστικές αλλά και τις μη εκτελεστικές ε, θέσεις. Δηλαδή, για μας θα πρέπει να αφορά και τους εκτελεστικούς διευθυντές και ε, τα στελέχη. Απλώς οι στόχοι είναι διαφορετικοί. Η πιο σημαντική αλλαγή που κάναμε είναι ε, ότι θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας μια ποικιλία διαδικασιών επιλογής. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασικά η βάση είναι η διαδικασία για τους κανονικούς υπαλλήλους, τα στελέχη, ε, όχι όμως τα διευθυντικά στελέχη. Ε, υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία εκεί στους διορισμούς, ε, έχουν εκλογές άλλες φορές, ε, λαμβάνουν υπόψη και άλλα κριτήρια ε, τα προσόντα, την εμπειρία, την εθνικότητα, ε, την ε, εκπροσώπηση, αντιπροσωπευτικότητα και όλα αυτά. Δεν είναι η συνήθις διαδικασία επιλογής προσωπικού. Και είπαμε, βεβαίως θα πρέπει οι εταιρείε να προσαρμόσουν τις διαδικασίες και να στοχεύουν το 40% του φύλου που υποεκπροσωπείται. Αλλά τα αφήνουν στα χέρια των κρατών μελών όσο και των επιχειρήσεων να αποφασίσουν πώς θα τα ρυθμίσουν αυτά δεν τους βάζουν κανένα κορσέ. Αλλά άλλο που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να εστιάσουμε στη σύνολη διαδικασία επιλογής προσωπικού και προσλήψεων. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής εστιάζει στο τελικό στάδιο, όπου έχει γίνει ένα σύντομος κατάλογος ε, shortlist ε, των ε, υποψηφίων και πρέπει να γίνει τελική επιλογή. Ωραία. Εμείς τι λέγουμε εκεί. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει μια πλειάδα υποψηφίων και αν δεν υπάρχει γυναίκα με ίδια προσόντα ή περισσότερα, τότε προφανώς δεν πρόκειται να επιλεγεί. Αν μια εταιρεία δεν επιλέγει από το υποεκπροσωπούμενο φύλλο, δεν, ε, ε, ε, θα πρέπει να αναφέρει γιατί δεν έγινε αυτό, πώς επέλεξαν την τελική ομάδα υποψηφίων κτλ. Υπάρχει υποχρέωση δηλαδή αναφοράς αλλά και εξήγηση. και προσπαθήσαμε να κάνουμε μια διάκριση εκεί. Ε, από τη μια εταιρείε που έχουν καλές επιδόσεις και έχουν προσαρμόσει τις διαδικασίες Λοιπόν, να γίνει μια διάκριση μεταξύ των καλών μαθητών και των κακών μαθητών. Οι καλέ εταιρείε που έχουν τι καλέ διαδικασίε απλώ θα δίνουν τα στοιχεία στι αιτήσει εκθέσει, δεν θα είναι υποχρεωμένε να δηλώνουν ένα σωρό στοιχεία. Από την άλλη, εκείνοι που έχουν ακόμα κακέ επιδόσει και κυριαρχεί το ένα φύλλο, έχουν πιο βαριέ υποχρεώσει αναφορά και εξηγήσεων. Ε, Λεπτομερώ θα πρέπει να δικαιολογούνται, να απολογούνται γιατί συνέβησαν όλα αυτά, πώ φτάσαμε εδώ και τι πρέπει να αλλάξει στο μέλλον. Uh, Στη συνέχεια. Ε, ήταν λίγο ασαφής η διατύπωση ως προς την εφαρμογή. Γενικά εμείς είμαστε υπέρ της ρήτρα αναστολής. Αν ένα κράτος μέλος έχει μέτρα, τα οποιαδήποτε μέτρα που προβλέψει, ε, θα πρέπει να ελέγχει τη λειτουργία τους. Εάν τα κράτη-μέλη εμπιστεύονται τα εθελοντικά μέτρα, καλή τους τύχη και για τους με χαρά τους, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να αξιολογούν αν λειτουργούν αυτά. Σε αντίθετη περίπτωση, μέχρι το 2017 προτείναμε να τεθεί σε ισχύ αυτόματα η οδηγία και να αρχίσουν οι προσαρμογές. Και ένα τελευταίο σχόλιο Είπαμε, αρμόδιε επί τη ουσία επιτροπές είναι Γιούρι και ΦΑΜ, γυναικών και νομικών υποθέσεων. Παρέτειναν την προθεσμία του και μπορούμε και εμεί να την παρατείνουμε, γιατί κανονικά τώρα προβλέπεται μέσω μετά την τυρκουά εβδομάδα. Δεν έχει πολύ χρόνο ο κόσμο να σκεφτεί και να κάνει τροπολογίε. Οπότε, προτείνουμε να παραταθεί η προθεσμία ε, κατάθεση τροπολογιών αλλά και ο χρόνος που θα έχουμε για να ψηφίσουμε. Επίσης, ευχαριστώ. Vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν ζητήσει το λόγο βεβαίως οι σκιώδεις, οι συγγήτριες και οι συγγητές. Η κυρία ούτε πρώτη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δέχομαι την πρόταση της Κομισιόν και χαίρομαι ιδιαίτερα για το σχέδιο οδηγίας. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί η εξισορρόπηση των φύλων σε διάφορους τομείς, όπως και στα διοικητικά συμβούλια εταιριών. Η εισηγήτρια κυρία Κορνέλισεν μας παρουσιάζει μία πολύ σοβαρή γνωμοδότηση και πιστεύω ότι η πρόταση διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογή πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τα μη διοικητικά στελέχη αλλά και τα διοικητικά. Επίσης συμφωνώ για την ποικιλότητα των διαδικασιών επιλογής, δηλαδή την τροπολογία 23 γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη μπορεί να ακολουθούν διαφορετικές διαδικασίες για την επιλογή εκπροσώπων του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα για τις κυρώσεις. 34, 35 και 36, τροπολογίες 34, 35 και 36, συμφωνώ ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές. Αλλά και όμως Πρέπει επίσης να συζητήσουμε περισσότερο την πρόταση της εισηγήτριας για τον περιορισμό της χρηματοδότησης της ενοκής χρηματοδότησης από, για εταιρείε που δεν σέβονται την οδηγία. Επίσης πρέπει να συζητήσουμε πιο λεπτομεριακά πώς θα εφαρμοστούν τα κίνητρα που προτείνονται για διαδικασίες δημοσίων προμηθειών. Έχω λοιπόν μερικές αμφιβολίες και προτάσεις για τις κυρώσεις και απορίες ως προς τη χρημα... ενωσιακή χρηματοδότηση και για τις δημόσιες πραμήθειες. Τώρα για τις τροπολογίες 17 και 28 που αναρωτιόσασταν. Λοιπόν, η ιδέα η ίδια που εκφράζουν είναι καλή, αλλά πρέπει να προβλεφθεί και η δυνατότητα χορήγησης κινήτρων από τα κράτη σε εταιρείε για την καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας εφόσον οι εταιρείε διαπιστώσουν ότι δεν ακολουθήθηκαν οι νενομισμένες διαδικασίες επιλογής ιδιαίτερα ως προς την εξισορρόπηση των φύλων. Αν υπάρχει μια τεράστια κατασκευαστική εταιρεία κυρίως ανδρών δεν σημαίνει αυτό ότι απαγορεύεται στις γυναίκες να μπουν στο διοικητικό της συμβούλιο, αλλά θα έπρεπε να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος διατύπωσης της οδηγίας ώστε η πρόταση να είναι ακόμη πιο αποτελεσματική. Τέλος, όπως είπε η κυρία Κορνέλισεν, υπάρχουν αρκετές διχογνωμίες και πάθη γύρω από αυτή την πρόταση. Τα περισσότερα κράτη δέχονται μεν την πρόταση, αλλά θα ήθελα να φτάσουμε στο, σε ένα τελικό αποτέλεσμα που να είναι αποδεκτό από όλους και όλες. Να αναζητήσουμε δηλαδή συμβιβασμούς και συνενέσεις ώστε η οδηγία αυτή να μην μπλοκαριστεί για χρόνια και χρόνια στο Συμβούλιο όπως έχει γίνει με άλλες. Και καλό θα ήταν να καταφέρουμε να την εγκρίνουμε κατά αυτήν τη θητεία. Μάλιστα. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με αυτό το τελευταίο. Διότι θα πρέπει να έχουμε και κάτι να προτείνουμε στην προεκλογική εκστρατεία. Κυρία Μπάουερ, επόμενη, παρακαλώ. So, I would like to support the... Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να στήριξω την πρόταση της κυρίας Κορνέλισεν όσον αφορά την παράταση της προθεσμίας υποβολής τροπολογιών, γιατί ε, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών έχει αλλάξει το δικό της το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την έγκριση της ε, οδηγίας αυτής, της έκθεσης για την οδηγία. Εκτιμώ ιδιαίτερα την εργασία που έχει κάνει η συγγήτρια για την πρόταση αυτή. και έχω και εγώ κάποια ερωτήματα και κάποιες αφιβολίες. Και ενδεχομένω θα μπορούσα να κάνω και κάποιες προτάσεις ε, τροποποιητικές. Καταρχάς πιστεύω ότι θα ήταν αναγκαίο να διασαφηνίσουμε τη νομική βάση. Έχουν διεξαχθεί κάποιες συζητήσεις στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων όσον αφορά την ε, νομική βάση. Και αυτός είναι μάλλον ο βασικός λόγος για τον οποίο αναβλήθηκε κάπως η όλη διαδικασία. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά το ζήτημα της νομικής βάσης. Έχω επίσης την εντύπωση ότι η πρόταση της Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ καλά ισορροπημένη. Και δεν ξέρω βέβαια αν θα τα καταφέρουμε. Εγώ πάντως ε, ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε μία λογική διάρθρωση σε αυτήν την ε, πρόταση. Γιατί ξέρετε βέβαια ότι μπορούμε να έχουμε πολλές διαφορετικές ιδέες, ωστόσο η βασική προϋπόθεση είναι να δούμε αν ε, μπορεί να γίνει αποδεχθή η πρόταση αυτή από το Συμβούλιο. Και εγώ αυτή τη στιγμή έχω κάποιες ε, αμφιβολίες ως προς αυτό. Προφανώς όμως θα προσπαθήσουμε να επεκτείνουμε είτε το πεδίο εφαρμογής είτε τις κυρώσεις που προβλέπονται σε αυτή την πρόταση. Για παράδειγμα, Όσον αφορά την τροπολογία 28, πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη. Γιατί πραγματικά το να επιβάλλουμε την πρόταση αυτή σε διάφορους τομείς όπου δεν υπάρχουν τελικά, δεν απασχολούνται γυναίκες, κάτι τέτοιο θα ήταν απαράδεκτο. Όσον αφορά τώρα τις κυρώσεις, Έχω αρκετέ αμφιβολίε όσον αφορά τι κυρώσει και τι κυρώσει που είχαμε προβλέψει παλαιότερα όσον αφορά το gender pay gap, τη διαφορά δηλαδή στην αμοιβή ανδρών και γυναικών. Νομίζω ότι οι κυρώσει τουλάχιστον που είχαν προβλεφθεί θα ήταν πολύ πιο χρήσιμε σε αυτή την περίπτωση, όταν υπάρχει διαφορά αμοιβή, διαφορά μισθού μεταξύ ανδρών και γυναικών, παρά εδώ, παρά στο συγκεκριμένη αυτή πρόταση. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Κάθε φορά προσπαθούμε να επεκτείνουμε το πεδίο αυτών των κυρώσεων, ιδίω όσον αφορά αυτά τα μη. Μάλλον, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την επέκταση τη πρόταση στα εκτελεστικά διοικητικά στελέχη. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ε, να αποφύγουμε να αποτύχουμε την πρόταση αυτή όπως έγινε με την πρόταση για την ε, άδεια μητρότητας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο και να αποτύχουμε την πρόταση αυτή θα στείλουμε ένα πολύ αρνητικό μήνυμα Ή δεν θα καταφέρουμε τελικά να προωθήσουμε τα σημεία τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε την πρόταση αυτή. Και βέβαια προσβλέπω σε μια επικοδομητική συνεργασία για να βρεθεί και μια κοινώ αποδεκτή λύση. Ευχαριστώ, κυρία Χάρτη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Συμφωνώ με τις περισσότερε από τι προτάσει που κάνει στη γνωμοδότησή τη. Καταρχάς να σας πω ότι υποστηρίζω προφανώς την ίδια την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είδαμε ότι σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν κάποιες ε, σχετικές πρωτοβουλίες με αυτορύθμιση, με μη δεσμευτικά μέτρα και οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν αποδώσει τελικά. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ασχολείται με τα μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη. Η συγγήτρια μας λέει η πρόταση να ισχύει πλέον και για τα εκτελεστικά διοικητικά στελέχη. Συμφωνώ με την πρόταση αυτή. και είναι πολύ σημαντικό και τα ίδια τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να υπόκεινται στις ίδιες ποσοστώσεις φύλου. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε περαιτέρω, πιστεύω. Συμφωνώ επίσης με την πρόταση της συγγήτριας ότι θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη και στις εταιρείε να έχουν ένα κάποιο βαθμό ευελιξίας για το πώς θα καταφέρουν να προσαρμόσουν τη διαδικασία επιλογής νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στα αποτελέσματα και θα πρέπει να αποδεχθούμε το ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά συστήματα επιλογή στα κράτη-μέλη. Ακούσαμε επίση διάφορε παρατηρήσει από του συναδέλφου για το ζήτημα της διασφάλισης της πρότασης αυτής όσον αφορά το Συμβούλιο. Πιστεύω ότι θα πρέπει όντως να προωθήσουμε την προσέγγιση αυτή. Όσον αφορά τροπολογία 16, Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε αποκλεισμό από ε, κοινοτική χρηματοδότηση, περιορισμένη κοινοτική χρηματοδότηση. Δεν συμφωνώ ούτε με τα δύο τμήματα της τροπολογίας αυτής. Ξέρετε ότι δεν συμφωνώ με το ζήτημα των μακροοικονομικών προϋποθέσεων και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να προβλέπετε κάτι τέτοιο σε αυτή την τροπολογία. Το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 16 αναφέρεται στην ε, επιλογή των εταιριών που μπορούν να συμμετέχουν σε δημόσιες συμβάνσεις. Και πάλι δεν είμαι καθόλου πεπισμένη θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε τα όσα λέγονται στην τροπολογία αυτή και δεν ξέρω αν θα ήταν και ευκταίο τελικά να γίνεται κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε ακόμα περισσότερο με την, με την εισηγήτρια. Συμφωνώ με τις τροπολογίες 26 και 31 για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών και άκουσα τα όσα είπε η κυρία Μπάουερ για τη νομική βάση. Προφανώ χρειαζόμαστε εδώ μεγαλύτερη σαφήνεια και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε μια πιο σαφή νομική βάση τι επόμενε εβδομάδε. Άρα είναι καλό το ότι έχουμε παρατείνει την ημερομηνία υποβολή των τροπολογιών. Και πρέπει να δούμε και ποια θα είναι η θέση του Συμβουλίου. Εμεί βέβαια εδώ είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε τη δική μα τοποθέτηση, αλλά παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια κάποια συμφωνία για την πρόταση αυτή με το Συμβούλιο. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτή τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στα δυο μας θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χάρκιν. Και τώρα ο κύριος Μπένιον. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ σύντομα εγώ μόνο. Εγώ γενικά είμαι κατά των ποσοστώσεων, πόσο μάλλον εδώ όπου αναφύονται ποσοστώσεις, εγώ είμαι αντίθετος. Είναι μηχανιστική αντίληψη αυτή και προσέγγιση. Και δεν προσφέρεται σε καμία ε, δραστηριότητα της ζωής. Συμφωνώ όμω εδώ με την κυρία Κορνέλησεν σε ένα σημείο. Τώρα έχει γίνει κάποια δουλειά για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής των στελεχών. οι αντικρουόμενες ε, προτεραιότητες αρχίζουν σιγά σιγά και ξεδιπλώνονται. Και είναι πολύ δύσκολο με νομική βάση να βρεθεί μια υποστήριξη σε ένα πολύ άκαμπτο σύστημα ποσοστώσεων. Ποιο είναι το ζήτημα τώρα, από ό,τι μπόρεσα εγώ να καταλάβω. Κινείται περισσότερο προς πιο ισόρροπες ε, ε, επιλογές τελικών καταλόγων shortlist μερικών υποψηφίων και ορισμένοι να απολογούνται ή να δικαιολογούνται γιατί το πράττουν αυτό. Ε, αυτό είναι κάτι που μπορώ να δεχτώ, έστω και με βαριά χάρια. Οι θέσεις των διευθυντών δεν έρχονται μαζικά μία-μία ελευθερώνονται. Άμα έχει πάρα πολύ σκληρή ποσόστοση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιλέξει προσωπικό. Γιατί θα πρέπει να γίνει φωτογραφική διάταξη εκ των προτέρων, πράγμα παράνομο. Με ενθάρρυνα λοιπόν αυτά που άκουσα. Θα μελετήσω βέβαια σε λεπτομέρειες την πρόταση, αλλά μάλλον φαίνεται ότι καλά το πηγαίνει. Η κυρία Κορνέλησεν προς μια πρόταση που θα μπορούσα μέχρι και εγώ να υποστηρίξω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δύο μου είπαν ότι είναι εκπρόσωποι. Ο κύριος Κόντικ και ο κυρία Σότ από τη Γενική Διεύθυνση Just. Ποιος θέλει να αρχίσει. Παρακαλώ. Ε, Όχι, η κυρία Σρότ απουσιάζει. Εγώ είμαι ο Μιχαήλ Γκρόντεκ. που εργάζομαι ως νομικός στην Γενική Διεύθυνση Justice. Για το νομικό υπόβαθρο να πω δύο λόγια. Η Κομισιόν είναι απολύτως πεπισμένη ότι το άρθρο 157.3 είναι η σωστή νομική βάση, το σωστό νομικό υπόβαθρο για την ισότητα των φύλων που αναγνωρίζεται και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι αφορά εργαζόμενους και άλλους. Α, και τους ε, αυτοαπασχολούμενους. <clears throat> Παραδείγματος χάρη στην περίπτωση Ντανόσα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων εταιριών πρίμα φάκη πληρούν τις συνθήκες για να θεωρηθούν αυτοαπασχολούμενοι. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να επαναλάβω να... ότι η Κομισιόν είναι πεπισμένη ότι μπορούν να γίνουν πολλά θετικά με βάση εκείνο το άρθρο που σας έλεγα. Και το σημείο 1, το άρθρο 1 της οδηγίας που λέει ότι ο στόχος της είναι και η επιταχυμένη πρόοδος για την ισότητα των φύλων αλλά και επαρκή χρόνο για ελαστικότητα για τις εταιρείε για να εφαρμόσουν τον νόμο αυτόν. Το άρθρο λοιπόν εκείνο μας αρέσει και αναμένουμε τις τροπολογίες για να δούμε αν θα πληρωθούν και οι δύο αυτοί όροι και πρόοδος και φιλικότητα προς τα επιχειρήσεις. Ευχαριστώ και η συγγήτρια για να κλείσει. Παρακαλώ να συνοψίσετε για να απαντήσετε και σε πολλές ερωτήσεις που σας έγιναν. Καλώς, ευχαριστώ πολύ κύριε Κορνέλισεν. Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας. Χαίρομαι που βλέπω τέτοια μεγάλη υποστήριξη Πολλές ε, ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν βέβαια και επί της ουσίας, αλλά και επί της θέσης του Συμβουλίου οπωσδήποτε, γιατί συμφωνώ με όλους όσοι είπαν ότι χρειαζόμαστε πραγματικά. Μεγάλη προθυμία και πνεύμα συμβιβασμού για να, γίνει αυτό πραγματικότητα και για τις γυναίκες αλλά και για τους άνδρες. Να μην παραμείνουν αυτά στα χαρτιά σε ένα ράφι, σε ένα σερτάρι του Συμβουλίου προς απόφαση κάποια στιγμή. Σύντομα να απαντήσω σε μερικά από τα σχόλια που κάνατε για τον κύριο Μπάνι. Πιστεύω ότι όντως έχουμε κινηθεί πολύ προς τη δική σας κατεύθυνση. Δεν είναι θέμα ποσοστώσεων. Ούτε επιβάλλουμε αριθμό γυναικών που θα πρέπει να συμμετέχουν ή να διορίζονται στα διοικητικά συμβούλια στόχους θέλουμε να θέτουν οι εταιρείε και διαδικασίες να προσαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε οι στόχοι αυτοί να μπορούν να υλοποιούνται. Λαμβάνονται υπόψη όμως και δεχόμενοι αντικειμενικοί λόγοι που απαγορεύουν κάτι τέτοιο καμιά φορά. Ως ε, για τις κυρώσεις αυτές αφορούν τις εταιρείε που δεν κάνουν καμία προσπάθεια να προσαρμοστούν. όχι το αποτέλεσμα δηλαδή, το θέμα είναι η πρόθεση, αυτό μας ενδιαφέρει. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν κυρώσεις είτε για εκείνους που αδρανούν είτε για εκείνους που δεν μπορούν να εξηγήσουν γιατί δεν έχουν ε, πετύχει τίποτα. Βεβαίως εργαζόμαστε πολύ σκληρά και οι νομικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου ε, για τον τρόπο αξιολόγηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια νομική εκτίμηση που λέγει ότι είναι εντάξει η νομική βάση. Την περασμένη εβδομάδα ήρθε η νομική υπηρεσία του Συμβούλου και λέει ότι δεν είναι εντάξει. Και τώρα εμείς είμαστε το τρίτο θεσμικό όργανο και το σημαντικότερο δεν λέω και θα πρέπει να περιμένουμε και τη δική μας νομοδότηση. Θα τα κοιτάξουμε. Ε, ελπίζω πριν τη λήξη της προθεσμίας θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε σε μεγαλύτερο βάθος. Έτσι και τώρα παρατάθηκε η προθεσμία και μας δίνει κάποιο χρονικό περιθώριο. Τώρα το θέμα των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών σε σχέση με τα εκτελεστικά. Ε, κοιτάξτε, εμεί δεν θέλουμε να ξεχυλώσουμε το πεδίο εφαρμογής. Ε, και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με τα εκτελεστικά στελέχη. Καλά, σε μία παράγραφο, μην νομίζετε κιόλα. Και τονίζουν σε όλες τις άλλες παραγράφους ότι πρόκειται μόνο για μία εκτελεστικά διοικητικά στελέχη. Δεν θα πρέπει να ε, διευρύνουμε λοιπόν το πεδίο εφαρμογής, απλώς να πούμε ότι αφορά και τα εκτελεστικά στελέχη, διότι ακριβώ σε επίπεδο εκτελεστικών στελεχών ο αριθμός των γυναικών η κυρία Μπλίνκεβιτσούτε αναφέρθηκε στην τροπολογία παριθμών 28. Ε, αυτό αφορά εταιρείε ε, που οι γυναίκε ή το υποεκπροσωπούμενο φύλλο είναι κάτω του 10% των εργαζομένων. Να εξαιρεθούν αυτές, λέγει. Μα Δεν καταλαβαίνω γιατί θέλει ε, να διαγραφεί αυτό. Ε, γιατί δεν μπορεί μια γυναίκα να είναι επικεφαλή σε μια χαλιβουργία. Μπορεί. Μπορεί. Δεν ξέρω, πέρασε από το Συμβούλιο, δεν έχω πρόβλημα. Αυτά νομίζω είναι τα περισσότερα. Για τις κυρώσεις Υπάρχουν παραδείγματα ε, σε κράτη-μέλη που επιβάλλουν κυρώσεις. Ας πούμε, αποκλείουν τις εταιρείε από συμμετοχές σε διαγωνισμούς ή τις περιορίζουν ή τη χρηματοδότηση. Πρέπει όμως να σας πω ότι οι κυρώσεις δεν εφαρμόζονται όταν οι εταιρείε δεν έχουν 40% γυναικών στα διοικητικά του συμβούλια. Δεν είναι αυτή η κύρωση. Η κύρωση επιβάλλεται στην εταιρεία που δεν κάνει προσπάθεια να εμπλέξει περισσότερες γυναίκες. Όχι σε αυτή που δεν πετυχαίνει το στόχο. Αυτά. Είμαι στη διάθεσή σας πάντα. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ερχόμαστε τώρα στο νέο χρονοδιάγραμμα και τη νέα προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών που είναι η 15η Μαΐου, 12 το μεσημέρι. Εντάξει, νέα προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 15 Πέμπτου 12 η μεσημερινή. Θα συζητήσουμε μετά αυτές τις τροπολογίες της συνεδρίαση της 19ης και 20ης Ιουνίου και στην Ολομέλεια. Όχι, προηγουμένως στις 9 Ιουλίου θα τις ψηφίσουμε και θεωρούμε ότι το Σεπτέμβριο θα εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλης. Αυτό είναι το νέο χρονοδιάγραμμα πλέον. Ωραία. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή και θα παραδώσω τώρα την Προεδρία στη συνάδελφό μου Νάντια Χίρσου. Λοιπόν, καλημέρα σας και από δική μου πλευράς. Ευχαριστώ πολύ Ελίζα Μπέτ που ανέλαβε την Προεδρία. Ερχόμαστε στο σημείο 15 τώρα, σχεδιασμό λέει τη εκπαίδευση. Έχουμε την γνωμοδότηση της κυρίας Κίνγκα Γκέρνς να συζητήσουμε και Παρακαλώ την κυρία Γκιόνς να μας ε, παρουσιάσει τη γνωμοδότησή της. Σε ευχαριστώ Νάντια. Η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Πολιτισμού και η Κατερίνα Μνταμπάλοβα είναι η εισηγήτρια. Η δική μας επιτροπή συντάσσει μια γνωμοδότηση. Προσπαθήσαμε να συντάξουμε μια γνωμοδότηση που να καλύπτει όλες τις πτυχές της πρότασης και κυρίως πτυχές που είναι σημαντικές για τη δική μας την Επιτροπή όσον αφορά την απασχολησιμότητα, όσον αφορά την προετοιμασία των νέων για την αγορά εργασίας, αλλά προσπαθούμε επίσης και να επικεντρωθούμε στην πτυχή της κοινωνικής ένταξης, δηλαδή να καταφέρουμε να ενσωματώσουμε αυτούς οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι ή που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Να τους προτιμάσουμε δηλαδή και αυτούς, να τους βοηθήσουμε να ενσωματωθούν στην κοινωνία, να καταφέρουν να ταχθούν επιτυχία στην αγορά εργασίας. Προσπαθούμε να αφαιρθούμε σε κάποιες ε, οριζόντιες δεξιότητες, στις οποίες αναφέρθηκε και η Επίτροπος Βασιλείου χθε. όσον αφορά δηλαδή σημεία όπως η ε, ενεργή συμμετοχή του πολίτη στα κοινά α, γλωσσικές δεξιότητες, δεξιότητες που έχουν να κάνουν με τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία κτλ. Και προσπαθούμε επίσης να έχουμε ένα σύστημα εκπαιδευτικό, το οποίο θα είναι ολοκληρωμένο και θα, δεν, δεν θα έχει κανένα αποκλεισμό και που ουσιαστικά θα εντάσει και κάποιες ασθενείς ομάδες, ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως η Ρωμά και άλλοι και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε επίση και το ζήτημα της πρόορης αποχώρησης από το σχολείο. Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα πρόληψης του φαινομένου αυτού και να προβλέψουμε και κάποιες εξωσχολικές δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές θα μπορούν να συμμετέχουν από πολύ τρυφερή ηλικία. Δεξιότητε που ουσιαστικά θα βοηθήσουν στη συνέχεια τα παιδιά να ενταχθούν καλύτερα όταν μεγαλώσουν στην αγορά εργασία. Θέλουμε επίση να έχουμε καλύτερη μετάβαση μεταξύ εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης, Θεωρούμε επίση ότι θα πρέπει όμως να προετοιμαστούν καταλήλω και οι καθηγητέ, να προβλέπονται προγράμματα κατάρτιση καθηγητών, να εξοικειωθούν με διαφορετικού πολιτισμού και να αναπροσαρμόσουν τελικά τα μαθήματά του ε, στου ε, τρόπου επικοινωνία και μάθηση των φοιτητών του. Είναι σύντομη η γνωμοδότηση, τουλάχιστον στην πρώτη σε αυτή μορφή, στο πρώτο σχέδιο γνωμοδότηση που έχουμε μπροστά μας. Προσβλέπω στις τροπολογίες που θα υποβάλλετε. Να σας πω απλώς ότι έχουμε λάβει γνωμοδοτήσεις από διάφορα Ινστιτούτα και οργανισμούς, από την Business Europe, από διάφορα ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγινε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση με αυτούς τους πολλούς διάφορους οργανισμούς, οι οποίοι ε, μοιράστηκαν μαζί μας την ε, άποψή τους. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να καταφέρουμε να ακούσουμε όλες αυτές τις απόψεις από τους διάφορους οργανισμούς ή τις εταιρείε. Και ουσιαστικά αυτό που υπόθηκε είναι ότι ε, η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντική για να πετύχουμε δύο βασικούς στόχους. Από τη μια την απασχολησιμότητα και από την άλλη μια ισορροπημένη ζωή ουσιαστικά. Ορισμένοι είπαν ότι θα πρέπει να μεταβάλουμε πολλά σημεία της πρότασης, άλλοι μας είπαν οι συνάδελφοι ότι η γνωμοδότηση αυτή αποτελεί μια πολύ καλή βάση και πρέπει να σας πω ότι σε μία εβδομάδα λίγη η προθεσμία στις 30 Απριλίου για την υποβολή τροπολογιών. Θα ήθελα και εγώ να υποβάλω κάποιες ε, τροπολογίες και δεν κατάφερα να καλύψω όλα τα σημεία που θέλω να καλύψω στη σύντομη αυτή γνωμοδότηση. Η ε, εξέταση των τροπολογιών προβλέπεται στα τέλη Μαΐου, στις 29 και 30 Μαΐου δηλαδή. Θα εγκρίνουμε τη γνωμοδότηση στις 19 Ιουνίου, στις 20 μάλλον Ιουνίου, θα ακολουθήσουμε έπειτα το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και θα εγκριθεί από την Επιτροπή Πολιτισμού η έκθεση αυτή το Σεπτέμβριο. Θα ασχοληθούν δηλαδή με το φάκελο αυτό λίγο αργότερα από εμά στην Επιτροπή Πολιτισμού. Πάντω είναι σημαντικό εμεί να καταφέρουμε να του δώσουμε την γνωμοδότησή μα το συντομότερο δυνατό. Αυτά είχα να πω εντάχει. Περιμένω τώρα να ακούσω τη γνώμη των υπολείπων συναδέλφων. Σε ευχαριστούμε, Κίνγκα. Ο Μπέκερ έχει λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια ως μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης. Είμαι και εγώ σκιώδης εισηγητής στην Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης για την έκθεση αυτή και θα ήθελα να σας πω και τη δική μου την άποψη. Χαιρετίζουμε την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, έρχεται την κατάλληλη χρονική στιγμή Δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή αν προωθείται ιδιαίτερα ή όχι το ζήτημα της καινοτομία. Νομίζω ότι θα πρέπει να δρομολογήσουμε τώρα την έκθεση αυτή, γιατί έχουμε ήδη μπροστά μας κάποιες πολύ σημαντικές προκλήσεις στο μέλλον. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με το ζήτημα των δεξιοτήτων, με το ζήτημα της απασχολησιμότητας των νέων, να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στο ζήτημα αυτό της απασχόλησης και συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι η πνευματική ολοκλήρωση επίσης των νέων είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν υπάρχει δηλαδή μια αντίθεση ανάμεσα στην πνευματική ολοκλήρωση και την απασχολησιμότητα. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθήσουμε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης, τυπική, επίσημη και άτυπη, η επαγγελματική κατάρτιση, η μαθητεία, οι ξεσχολικές αυτές δραστηριότητες, οι οποίες αναφέρθηκε η συγκήτρια, συμβάλλουν πάρα πολύ στην ε, περαιτέρω απασχολησιμότητα των νέων. Και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ε, ευνοϊκή ε, στάση. Επιτρέψτε μου να αφαιρθώ λίγο στις δικές μου τροπολογίες. Ομολογώ ότι δεν κατάλαβα πάρα πολύ τι σχέση έχει η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Δεν κατάλαβα πού κολλάει εδώ. Ίσως να φταίει η δική μου νοημοσύνη, αν το εξηγήσετε. επίσης, Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα θέμα ε, μικρό μεροληψίας. Ε, σωστά αναφέρονται εδώ οι Ρωμά, αλλά δεν πρόκειται για τους Ρωμά, για όλες τις μειονότητες. Νομίζω καλύτερα ε, μπορούμε να το πούμε ως γενική ρίση. Το θέμα των γλωσσικών δεξιοτήτων είναι από τα κυρίαρχα για μένα. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την προσχολική ηλικία και από πολύ νωρί με την εκπαίδευση των ε, παιδιών. Αυτές οι γλωσσικές δεξιότητες και ικανότητες είναι το κλειδί για την εκπαίδευση και την ε, μετεκπαίδευση και την κατάρτιση γενικότερα, παντού. Ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, που σπανίως ε, προσλαμβάνει τις σωστές διαστάσεις, είναι το να μαθαίνει κανείς πώς να μαθαίνει. Δηλαδή, ε, στα σχολικά προγράμματα δεν υπάρχει ένα ελάχιστο διδακτικής, δηλαδή να μπορεί ο μαθητής να καταλαβαίνει πώς θα μαθαίνει. Αυτό έχει να κάνει και με την ανάγνωση, αλλά και με τεχνικές εκμάθησης. Υπάρχουν πάρα πολλές άριστες, τις οποίες όμως εμείς δεν διδάσκουμε. Θα πρέπει να αρχίσουν τα παιδιά κάθε φορά από τον Αδάμ και την Εύα. Κρίμα είναι αυτό. Είναι βασικό εργαλείο της εκμάθησης tool στα αγγλικά. Αυτό αφορά όλους τους ενδιαφερομένους, όλους τους ενεχομένους, αλλά κυρίως τους μαθητές. Θα πρέπει να γνωρίζουν τη σύγχρονη τεχνολογία πληροφορίας και να τη διδάσκονται και θα πρέπει να μπορούμε να το απαιτούμε αυτό και από τους δασκάλους για να κλείσει έτσι αυτός ο κύκλος. Σας ευχαριστώ ε, για τη φιλόδοξη αυτή εργασία και θα συνεισφέρω και εγώ από πλευρά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Um, next. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συνάδελφος Κοσμάνοβα δεν είναι εδώ σήμερα, γι' αυτό την αντικαθιστώ εγώ. Πρώτον, συγχαίρει την εισηγήτρια κυρία Γκόντς για το σχέδιο γνωμοδότησης που θεωρεί σημαντική βάση για τη μελλοντική μας συνεργασία. Πρώτος στόχος της στρατηγικής 2020 είναι να αυξηθεί ο ρυθμός απασχόλησης κατά 25%. στο στόχη, η μείωση του ρυθμού εγκατάλειψης του σχολείου και βελτίωση της ανώτερης παιδείας. Η βελτίωση της παιδείας θα αποτελέσει προώθηση και της οικονομίας γενικότερα και πρέπει να θεωρείται ε, και πρέπει να επιτυχάνεται με τρόπο όσο πιο ισότιμο και ισόνομο γίνεται. Επίσης πρέπει να κάνουμε τα σχολεία πιο ελκυστικά και τα εκπαιδευτικά προγράμματα να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών αλλά και της κοινωνίας οικονομίας. Αυτό αφορά και τις μειονότητες και τους μετανάστες. Το θέμα αφορά επίσης τις ευκαιρίες που έχουν οι μαθητές στην ανώτερη παιδεία, τους οποίους πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο λιτότητος. Εκείνη λέει μειώσεων, εγώ νομίζω εννοεί λιτότητας. Πρέπει να χορηγούνται πιο εύκολα μαθητικά και φοιτητικά δάνεια. Άλλη σύνδεση μεταξύ ανάπτυξης και παιδείας είναι η σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας. με συνεργασία των πανεπιστημίων, με οργανώσεις εργοδοτών κλπ. Και πρέπει να ενθαρρύνουμε τους διδάσκοντες οι οποίοι Κατά την τελευταία μελέτη που έγινε το 12 για την παιδεία, δεν έλκονται και τόσο πολύ στον τομέα αυτών εργασίας. Καταληκτικά, ίσως να ήταν χρήσιμο να προωθηθούν όλες οι δυνατότητες που δίνονται για χρηματοδότηση της παιδείας στην Ένωση, ιδίως για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Thank you, Marian. Ευχαριστούμε Μαριάν. Μήπως κανείς από την Κομισιόν θέλει να πει τίποτα εσείς εκεί κάτω. Ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Κλαβδία Τσερνιλόγκα. Είμαι από την Κομισιόν και την Υπηρεσία της Παιδείας. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή και την εισηγήτρια για το σχέδιο αυτογνωμοδότησης που είναι πολύ συνοπτική και συγκεκριμένη και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη για μεγαλύτερη περισσότερη επένδυση στην παιδεία γιατί πάντοτε έχει θετικά αποτελέσματα. Επίσης η ε, απόκτηση οριζοντίων δεξιοτήτων είναι κάτι που θέλω να τονίσω ιδιαίτερα γιατί βελτιώνει την απασχολησιμότητα αλλά και την αυτονομία των νέων και η σύνδεση βέβαια μεταξύ παιδείας και αργότερης εργασίας. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι τον Ιούλιο θα αρχίσουμε ένα πρόγραμμα δημιουργίας συμμαχιών και εταιρικών σχέσεων για μαθητεία ώστε οι εργοδότες να προσφέρουν μεγαλύτερες, περισσότερες εμπειρίες σε νέους. Τέλος, σας ευχαριστώ που σημειώνετε και τη σημασία που έχει η επένδυση στους διδάσκοντας και διδάσκουσες. Πρέπει να βοηθηθούν και αυτοί γιατί αντιμετωπίζουν συνεχώς καινούργιες απαιτήσει και πρέπει να αποκτούν όλο και καινούργιες δεξιότητες Άρα η συνεχής επιμόρφωση είναι σημαντική, αλλά επίσης πρέπει να τη διατηρήσουμε την ελκυστικότητα του επαγγέλματος του καθηγητή. Ευχαριστώ πολύ και της καθηγητρίας. Ευχαριστώ. Ξαναδίνουμε το λόγο στην συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκένς. Ε, σας ευχαριστώ επίσης για τα σχόλιά σας. Εγώ αυτό που προσπάθησε ναι, να γίνει όσο γίνεται πιο συνεκτική η γνωμοδότηση και ευσύνοπτη. Θα δούμε τώρα και με τις ε, τροπολογίες. Σκιώδης εισηγητής, ε, ο κύριος Μπέκερ είπε ότι είναι και στην Επιτροπή Πολιτισμού και χαίρομαι γι' αυτό. Θα υπάρχει έτσι καλύτερος συντονισμός. Κάνουμε και ε, συζήτηση αργότερα θα γίνει αυτή για την ενεργή συμμετοχή του πολίτη, για τις μειονότητες κτλ. Μα αυτό είναι από το βασικότερα για την ένταξη στην κοινωνία. Κυρίως των νέων που ενδεχομένως να κινδυνεύουν να αποχωρούν από τα σχολεία ή να αποκλείονται κοινωνικά. Αυτό είναι άλλη συζήτηση, όμως θα την κάνουμε αργότερα. Τα ίδια ισχύουν για τις μειονότητες, μετανάστες ανθρώπους με αναπηρίες νέους που χρειάζονται βοήθεια. Αλλά όλα αυτά δεν είναι του παρόντος, θα τα συζητήσουμε αργότερα. Και πραγματικά χρειάζονται πλαισίωση και βοήθεια όλοι αυτοί για να μπορέσουν να βρουν ε, στη συνέχεια δουλειά και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ και τη Μάριον Χάρκιν που τονίζει ότι δεν θα πρέπει να είναι μόνο προσβάσιμη αλλά και ελκυστική η εκπαίδευση. και να είναι ελκυστική και για ε, παιδιά που είναι από μεσαίες τάξεις, αλλά και παιδιά από άλλα στρώματα που ε, δεν πάνε και τόσο ε, πρόθυμα στο σχολείο. Η κρίση έχει επηρεάσει πάρα πολύ τις οικονομικές δυνατότητες των οικογενειών, αλλά και των σχολείων. Θέλω να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι προσπαθούμε να τονίσουμε το αυξημένο επίπεδο επενδύσεων. Ε, ναι, μπορεί να είναι κάτι που θα υπομιστούν από κοινού και ο ιδιωτικός τομέας και ο δημόσιος. Ναι, αλλά πώς θα γίνουν αυτές οι ΔΙΤ. Γιατί για μένα εκεί ακριβώς χρειάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση επένδυση. Επίσης, αυτονομία των νέων. είναι από τους βασικούς στόχους και καλή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών προφανώς όταν είναι σωστοί οι δάσκαλοι ε, κάνουν και καλή δουλειά. Ευχαριστώ, περιμένω να δω τις απολογίες σας και να συνεργαστώ μαζί σας. Ευχαριστώ. Thank you, King. Σε ευχαριστώ, Κίνγκα, η Πρόεδρος. Είπε ήδη ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, η προθεσμία 30 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι Συζήτηση των τροπολογιών 29 ή 30 Μαΐου. Συμβιβασμοί 19 Ιουνίου και στις 20 έγκριση στην Επιτροπή Απασχόλησης. We can go to the next point on the... Πάμε στο επόμενο θέμα στη μέση διάταξη. Κοινή συζήτηση είναι αυτή για τα θέματα 16 και 17, κανονισμός για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και το 17 είναι in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Είναι η πρώτη συζήτηση. Εμείς γνωμοδοτούμε στον κανονισμό του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σχετικά για το 16 και το 17. Δική μας συντάκτρια γνωμοδότηση είναι η κυρία Ντίτε Στρέλα. Στο σχέδιο γνωμοδότησης της έχει υποβάλει 14, 14 συγγνώμη, τροπολογίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και 8 τροπολογίες για τα διαγνωστικά, το 17 δηλαδή. Κυρία Στρέλα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η πρόταση αυτή είναι αποτέλεσμα ενός σκανδάλου με εμφυτεύματα στήθους, τα οποία ουσιαστικά προκάλεσαν πάρα πολλά προβλήματα σε πάρα πολλές γυναίκες στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και ουσιαστικά θέλουμε εδώ πέρα να υποστηρίξουμε περισσότερο τους ασθενείς και τους καταναλωτές, να καταφέρουμε να αφησίσουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στις ιατρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση. Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα τεχνικό και οι αρμοδιότητες Επιτροπής Απασχόλησης είναι ιδιαίτερα περιορισμένες στον τομέα αυτό. Συνεπώς η δική μας προσέγγιση είναι να βελτιώσουμε την ασφάλεια και την υγεία κάθε φορά που χρησιμοποιούν οι ιατρικές αυτές συσκευέ στους ασθενείς από, επαγγελματίε της υγείας. Θέλουμε ουσιαστικά να ενημερώσουμε κάποιες οδηγίες οι οποίες υφίστανται αυτή τη στιγμή, να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε επίσης στην τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο των τελευταίων ετών και να καταφέρουμε επίσης να αντιμετωπίσουμε και τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί εξαιτίας ε, των ε, ψεύτικων αυτών ε, εμφυτευμάτων στήθους που είχαν χρησιμοποιηθεί. Όπως λέγεται στην ιδεολογική σκέψη 71 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στόχος του κανονισμού είναι να εγγυηθούμε υψηλά επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας για τις ιατρικές συσκευές, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο υγείας και ασφάλειας και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των ασθενών, καθώς επίσης και των χρηστών και των υπόλοιπων ανθρώπων που έρχονται σε επαφή με τα ιατροτεχνολογικά αυτά προϊόντα. Στην παράγραφο 8 του παραρτήματος, αποσαφηνίζεται ότι οι ιατρικές συσκευές καθώς επίσης και οι διαδικασίες κατασκευής θα πρέπει να είναι τέτοιες έτσι ώστε να μειώνεται σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο ο κίνδυνος λίμωξης, μόλυνσης των ασθενών και των χρηστών των συσκευών αυτών. Επίσης, λέγεται ότι χρειαζόμαστε ιατρικές συσκευές οι οποίες θα είναι σε θέση να συμβάλλουν στο να μειώνεται ο κίνδυνος των ανθρώπων που τις χρησιμοποιούν. Οι ιατροτεχνολογικές συσκευές χρησιμοποιούνται κυρίως σε νοσοκομεία από επαγγελματίες της υγείας, αλλά χρησιμοποιούνται επίσης και σε άλλα περιβάλλοντα, όπως για παράδειγμα σε οίκους ευγυρίας ή ακόμη και σε φυλακές. Θέλουμε και στα περιβάλλοντα αυτά να προστατεύσουμε την ε, υγεία και την ασφάλεια των επαγγελματιών της υγείας, αλλά και όλων αυτών οι οποίοι εργάζονται σε βοηθητικά επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα απασχολούνται με, την, με τον καθαρισμό των συσκευών αυτών ή με την ε, αποκομιδή και διάθεσή τους. Αυτά είναι τα βασικά σημεία, βασικές προτεραιότητες της πρότασης αυτής. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ περισσότερο στον στόχο της ασφάλειας των συσκευών αυτών, καθώς επίσης και στο πώς μπορούμε να καταφέρουμε να συμβάλλουμε στο να δημιουργηθεί ένα πιο ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Και ουσιαστικά κατά αυτόν τον τρόπο η πρόταση αυτή συνδέεται με τις ε, υφιστάμενες οδηγίες που ήδη εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδίως με την Οδηγία 32-2010, σχετικά με την πρόληψη τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα στον νοσοκομιακό και υγειονομικό τομέα. Θέλουμε με την πρόταση αυτή να καταφέρουμε να μειώσουμε τα ποσοστά τραυματισμού και λίμωξης από τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Κάποια πολύ απλά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα επίδεσμοι ή ακόμα και ιδιαίτερα εξελιγμένα προϊόντα θα πρέπει να καλύπτονται από, το, από την πρόταση αυτή η οποία θα προστατεύει τόσο τους ασθενείς όσο και το, τους επαγγελματίε της υγείας. Χρειαζόμαστε συσκευέ που να ανταποκρίνονται σε όλα τα κριτήρια τα οποία θέτουμε και χρειαζόμαστε έναν σαφή, διαφανή κανονισμό που λαμβάνει υπόψη και την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο των τελευταίων ετών. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν περιλαμβάνονται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και λαμβάνονται υπόψη και στην πρόταση που έχει κάνει η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και λαμβάνονται υπόψη βέβαια και στο δικό μας το σχέδιο γνωμοδότησης για την Επιτροπή Απασχόλησης. Όσον αφορά την προθεσμία υποβολής τροπολογιών, η 25η Απριλίου είναι η προθεσμία και περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Ήδη ορισμένοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μου. Ορισμένοι μου είπαν ότι θα πρέπει να τονίσουμε περισσότερο τα σημεία που ασχολούν και δική μας την Επιτροπή Απασχόλησης στην γνωμοδότηση αυτή. Okay okay. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας. Η κυρία Χάρκιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και σας και την εισηγήτρια. Συμφωνώ απόλυτα ότι η υγεία και η ασφάλεια είναι σημαντικός στόχος της πρότασης αυτής και συμφωνώ επίσης ότι δεν πρέπει μόνο το προσωπικό της πρώτης γραμμής όπως οι γιατροί και οι νοσοκόμες να ενδιαφέρεται γι' αυτό αλλά και πιο απομακρυσμένο προσωπικό. Υποστηρίζω τις προτάσεις της λοιπόν στις τροπολογίες 5 και 8. Επίσης για υγεία και ασφάλεια λέει και συμφωνώ ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας πρέπει να προστατεύονται είτε με εμβόλια είτε με χρήση τεχνολογίας που να αποτρέπει τη βλάβη της υγείας τους και έχει και άλλες τροπολογίες όπως την 11 και τη 13 η εισηγήτρια και τις υποστηρίζω και αυτές. Έχω όμως και ένα ερώτημα για την ΕΠΤΑ. σύμφωνα με την Κομισιόν τα κράτη-μέλη συντονίζουν μεταξύ τους, ή μάλλον στο εσωτερικό τους, το θέμα της αναφοράς σοβαρών ατυχημάτων. Ενώ η Κομισιόν μας λέει ότι πρέπει να υπάρχουν και αναφορές άλλο, με άλλη μορφή από τη συνήθη. Από ό,τι διάβασα όμως, μου φαίνεται ότι η πρόταση στοχεύει στη δημιουργία μιας κεντρικής τραπέζης δεδομένων που να συνδυάζει διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα με, ένα ενιαίο, με μια ηλεκτρονική ενιαία υπογραφή. Να συνδυάζει δηλαδή όλα τα σχετικά στοιχεία. Ερωτώ λοιπόν την εισηγήτρια τι υπονοεί όταν τα λέει αυτά. Γιατί πολλαπλά συστήματα. Um, it's not just healthcare professionals. Επίσης δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι στο τομέα της υγείας και οι ασθενείς που πρέπει να αναφέρουν ε, τέτοια ατυχήματα. Report any suspected incidents at national level. Αλλά και οι carers που λέμε εμείς. Δεν ε, λέω τέτοια. και Ακριβώς ένας από τους λόγους που υπάρχει αυτή η οδηγία είναι και το σκάνδαλο των ΠΙΠ. Χρειάζεται λοιπόν πλήρη συντονισμό μεταξύ των χωρών μελών. Και τέλο προ προς την Κομισιόν, ένα θέμα ορισμού δηλαδή, πολύ συγκεκριμένο που δεν αφορά ακριβώς αυτή την έκθεση, ο ορισμός του τι είναι η ιατρική συσκευή. Σύμφωνα με τη σελίδα 29, μια ιατρική συσκευή μπορεί να είναι οτιδήποτε ελαφρύνει ή βελτιώνει κάπως τις επιπτώσεις μίας πληγής ας πούμε. Εγώ όμως θεωρώ ότι και μια Αναπηρική πολυθρόνα μπορεί να θεωρηθεί η ιατρική συσκευή. Όχι μόνο μηχανές δηλαδή. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Μάριον. Δεν βλέπω άλλο βουλευτή να ζητάει το λόγο. So I can give the floor to... Θα δώσω λοιπόν το λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Σπανού παρακαλώ. Ευχαριστώ. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, τους αξιότιμους βουλευτές που εργάζονται για αυτό το θέμα και την εισηγήτρια που ακριβώς ε, λέγει αυτό που εμείς περιμέναμε να ακούσουμε από την Επιτροπή σας. Ιδιαίτερα ε, αξιολογείται πάρα πολύ ψηλά την ασφάλεια και την υγιεινή συνεργασία και η δική σας Επιτροπή δίνει πάντα πολύ μεγάλο βάρος αυτά. είναι σημαντικά αυτά που μας λέτε σήμερα και χαίρομαι που ήδη ακούσαμε κάποια πρώτα σχόλια. Ε, ξέρετε, είναι και η πρώτη ευκαιρία ε, που το συζητούμε αυτό. Ε, έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε για πρώτη φορά τις απόψεις σας και είναι καλή η αρχή. Βλέπετε από τις δύο προτάσεις που καταθέσαμε ότι όλη η αντίληψη και όλη η φιλοσοφία πίσω από τις δύο αυτές ενισχυμένες προτάσεις είναι να ε, ενισχύσουμε την προστασία της ασφάλειας και της υγιεινής στην εργασία, όχι μόνο για τους ασθενείς, αλλά και για τους χρήστες ιατρικών συσκευών και τέτοιων προϊόντων, ιατροτεχνολογιών, αλλά και άλλα πρόσωπα που χειρίζονται τι συσκευέ αυτέ. Το είπε και η συγκήτρια, θα πρέπει να καλύπτονται ε, όλοι ε, όσοι έχουν σχέση με τη χρήση αυτών. Θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει ανάγκη να γίνονται διαβουλεύσεις με οργανώσεις επαγγελματιών της υγείας νοσηλευτών και ασθενών. Μα ήδη το πράττουμε αυτό, ήδη έχουμε διαβούλευση. Και να δούμε πώς θα ενταχθεί στην πρόταση αυτή. Είναι βασικό στοιχείο της λήψης αποφάσεων. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε στοχευμένη νομοθεσία, πρακτική που να μην δημιουργεί περαιτέρω προσκόμματα ή εμπόδια και να βελτιώνεται η ασφάλεια των ασθενών. Ήδη στις προτάσεις μας υπάρχει μια διάταξη και μια πρόνοια για τη συμμετοχή ε, των οργανώσεων στην υποομάδα, στην υποεπιτροπή που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Και εννοώ εδώ και τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς. Σε ό,τι αφορά την προσωπική ασφάλεια, την ασφάλεια του προσωπικού, η νομοθεσία θα πρέπει να τα σέβεται όλα αυτά που ισχύουν για τα ιατροτεχνικά προϊόντα και τις συσκευέ. Συμφωνούμε απολύτως με την αρχή αυτή και θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να εξετάσουμε ποιοι είναι οι καλύτεροι νομικοί τρόποι να ε, εξασφαλιστεί αυτό. Για τα δεοντολογικά θέματα, ε, στα κλινικά πειράματα ή επεμβατικές ε, κλινικές πρακτικές. Ξέρετε ότι αυτό το θέμα το συζητούμε ευρύτερα και για τα πειράματα, τις κλινικές δοκιμές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ευθυγραμμίσει, θα προσαρμόσει και την πρόταση αυτή σε ό,τι αποφασίσουμε με το συνομοθέτη. Γιατί γνωρίζετε ότι και ε, αυτό το θέμα ε, είναι υποδιαπραγμάτευση και στο Κοινοβούλιο. Τελειώνοντας, πριν απαντήσω στο ειδικό θέμα του ορισμού, Θέλω να πω ότι υπάρχει ανάγκη και εκεί χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας και την υποστήριξή σας να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις αυτές και να τελειώσουν, να ολοκληρωθούν. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό. Ε, διαβάζω στα έγγραφα της συζητήτριας και ακούω από την Επιτροπή σας ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η ασφάλεια και η υγιεινή συνεργασία θα πρέπει να εγκριθούν οι προτάσεις αυτές κατά τη διάρκεια της παρούσης θητείας και είναι προς όφελος όλων. Δράτω με λοιπόν τη σημερινή ευκαιρία για να σας ζητήσω την υποστήριξή σας. Και τέλος, για να έρθω στην ερώτησή σας για τον ορισμό, κυρία Χάρκιν. Να είναι ευρύς ο ορισμός, διότι καλύπτει και τα δύο στοιχεία που αναφέρετε. Αν υπάρχει κανένα θέμα γλωσσικό διατύπωσης, να το κοιτάξουμε. Αλλά η πρόθεσή μας είναι να συμπεριληφθούν ε, στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και οι συσκευές και ε, τα άλλα που είπατε. Ελπίζω να διευκρινίζει τη θέση μας. Αν έχετε ρωτήσει με χαρά να απαντήσουμε. Ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια. Καταπληκτική έκθεση, θαυμάσια, πολύ εύστοχη, πολύ ειδική και με χαρά να δούμε και τις απολογίες. Ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω το λόγο τώρα στην κυρία Στρέλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χάρκιν για την υποστήριξή της και για τις προτάσεις τις οποίες έκανε, οι οποίες ενδυναμώνουν τα όσα ήδη περιλαμβάνονται στις ε, προτινόμενες τροπολογίες. Όσον αφορά την τροπολογία 7 ιδιαιτέρως, που έχει να κάνει με τις ιατρικές συσκευέ. Λέγεται εδώ ότι τα κράτη-μέλη συντονίζουν τη δράση τους, διατηρούν ωστόσο άλλες μορφές εντύπων για την αφορά ύποπτων σοβαρών περιστατικών σε αρμόδιες εθνικές αρχές. Βέβαια ξέρετε ότι δεν έχουν όλοι οι πολίτες και όλοι οι χρήστες πρόσβαση στο διαδίκτυο και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε ορισμένες χώρες ισχύουν και διαφορετικές πρακτικές. Για παράδειγμα, τη διαδικασία υποβολής ε, παραπώνων για ορισμένες χώρες γίνεται διαφορετικά από ό,τι σε κάποιες άλλες. Διαφέρουν λοιπόν τα συστήματα καταγγελίας από τη μία χώρα στην άλλη. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς θα πρέπει εδώ πέρα να επιμείνουμε στην παραδοσιακή μέθοδο υποβολής ε, καταγγελίας ή παραπώνων και όντως θα πρέπει να έχουμε μια τυποποιημένες μορφές υποβολής καταγγελιών μέσω διαδικτύου. Όσα περισσότερα όμω μέσα έχουμε διαθέσιμα για τους πολίτες, όσο περισσότερη διαφορετική είναι οι διαθέσιμοι τρόποι υποβολή καταγγελιών, τόσο το καλύτερο τελικά, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να μείνουμε στον παραδοσιακό τρόπο. Όσον αφορά πάλι την τροπολογία 7, αλλά αυτή τη φορά για τον κανονισμό των in vitro διαγνωστικών ιατρικών συσκευών. Ως προς αυτό θα ήθελα να σας πω ότι ήδη υπάρχει μία πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπει διαβούλευση με τους συλλόγους των επαγγελματιών της υγείας και των νοσηλευτών. Νομίζω ότι θα μπορούσε κάτι τέτοιο να προβλέπεται και στο ίδιο το διατακτικό του κανονισμού. Κατά αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ενδυναμώνεται η παγιωμένη αυτή ε, τακτική διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν δεν κάνω λάθος, άλλωστε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνούν με τα σημεία αυτά. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους συναδέλφους μου για την υποστήριξή τους. Ευχαριστώ πολύ για τη συνηφορά σα και τα σχόλιά σας. Λοιπόν, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 25 Απριλίου στις 5 το απόγευμα, έγκριση στην Επιτροπή μας τον Ιούνιο. Ωραία. Τώρα επανερχόμαστε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Συζήτηση για τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής όσο αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχομένους από φυσικούς παράγοντες ηλεκτρομαγνητικά πεδία δηλαδή, η κυρία Μωρέν Σαρτιέ θα μας ενημερώσει για τη συμφωνία που επετεύθη από αυτού του θέματος στις 27 Μαρτίου με το Συμβούλιο στην πρώτη ανάγνωση. Η κυρία Μωρέν Σαρτιέ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, είδου ένα τριμερής διάλογος που μπορούμε να πούμε ότι μας γέμισε ικανοποίηση. Πάρα πολύ γρήγορα έκλεισε η συμφωνία. Πρέπει να σας πω σε μία συνεδρίαση τριμερούς διαλόγου καταφέραμε να συμφωνήσουμε με μία πρώτερη συντονιστική ε, προκατακτική συνεδρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες διότι ειλικρινά έχω πλήρη επίγνωση ότι η ποιότητα των δικών μας εργασιών εδώ μαζί με τις υπηρεσίες της Επιτροπής μας, τις οποίες και ευχαριστώ πάρα πολύ. Επί σειρά μηνών, ε, δεν ξέρω, 1,5-2 χρόνια συζητούμε αυτό το θέμα. Ε, όλες οι πολιτικές ομάδες και η διοίκηση καταφέραμε τελικά χάρη στη ε, ψήφο στην Επιτροπή να επιτύχουμε μια πάρα πολύ σαφή διαπραγματευτική εντολή επί της οποίας όλοι ήταν σύμφωνοι και τήρησαν τη γραμμή. Ήρθαμε λοιπόν ενωμένοι και ισχυροί στην τριμερή συνεδρίαση ε, μετά από έγκριση στην Επιτροπή μας στις 6 Δεκεμβρίου. Αυτή η νέα οδηγία θα θυμάστε έρχεται να διορθώσει εκείνη του 2004 η οποία δεν επέτρεπε πλέον να γίνονται διάφορες ιατρικές εξετάσεις βασικά θα απαγόρευε τη μαγνητική ε, τομογραφία. Είναι πάρα πολύ ισόρροπη λοιπόν η νέα ε, πρόταση με τις νέες διεθνείς οριακές τιμές. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό διότι η Ευρώπη ε, επέβαλε μια διεθνή εναρμόνιση για αυτά τα θέματα. Από την άλλη, η νέα οδηγία μας επιτρέπει προσωρινές παρεκκλήσεις, υπερβάσεις, τελείως ε, έκτακτες. Λαμβάνεται υπόψη βεβαίως πάντα η ασφάλεια και η υγιεινή των εργαζομένων, αλλά το όφελος από τη χρήση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων επίσης λαμβάνεται υπόψη. Λαμβάνουμε και τις προφυλάξεις μας διότι υποχρεώνουμε τους εργοδότες να αξιολογούν τον κίνδυνο εκ των προτέρων και να ενημερώνουν αντιστοίχως τους εργαζομένους. Δηλαδή, η νέα πλέον οδηγία επιτρέπει να χτίσουμε όχι μια νέα επιστήμη προφανώς, αλλά τα νέα επιστημονικά δεδομένα για να δούμε τι επιπτώσεις έχουν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στην υγεία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια νέα κατεύθυνση. Εκτίμηση κινδύνου. Μπορεί να δημοσιεύεται και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η οδηγία δεν εξετάζει τα μακροπρόθεσμα ε, αποτελέσματα, της επιπτώσεις, γιατί δεν τα γνωρίζουμε ακόμα. Αλλά υπάρχει δυνατότητα λοιπόν συλλογής ε, και με παρακολούθησης για να δούμε ποιες θα είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε περίπτωση που υπάρχουν αυτές θα είμαστε οι πρώτοι που θα ενημερωθούμε και θα καταθέσουμε νέα πρόταση για νομοθεσία. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι διότι όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν και είδαν τις θέσεις τους να αντανακλώνται στην πρόταση. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε Και επιπλέον, Είμαστε πάρα πολύ ακαμπτοί ως προς τη θέση σε ισχύ, την ημερομηνία δηλαδή για την έναρξη ισχύω της ε, οδηγίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιταχύνουμε τη μεταφορά στην αρχή προβλεπόταν μία τριετία από τη θέση σε ισχύ της οδηγίας να έχει μεταφερθεί σε εθνικό δίκαιο. Εμείς ζητήσαμε πρώτη προ... εβδόμου του 2016 να έχει μεταφερθεί σε όλες τις εθνικές νομοθεσίες. Την 1η Ιουλίου λοιπόν του 2016. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να εγκρίνουμε εμείς το συντομότερο τη δική μας θέση Αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ψηφίσει τον Ιούνιο του 2013 στην Ολομέλεια. Ε, Όλα τα διοικητικά μέτρα έχουν ληφθεί για να γίνει σε αυτή την Ολομέλεια η ψηφοφορία και στη συνέχεια το Συμβούλιο θα υιοθετήσει την άποψη του Κοινοβουλίου με στόχο να υπογραφεί η οδηγία από τους και ε, την 1η Ιουλίου του 2013 να δημοσιευθεί και στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εμείς τι θέλουμε να ψηφίσουμε σήμερα. Ε, euh, και ε, βάσει των νέων διατάξεων του άρθρου 70, είναι τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου, σας τηρούσαμε πάντα ενήμερους. Όλα αυτά που σας εξήγησα τώρα θα τα ψηφίσουμε το απόγευμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Ελίζαμπετ. Ο κύριος Σέρκας. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος της συναδέλφου Σιλβάνα Ράπτη, που είναι τώρα σε τριμερή διάλογο, ε, πρέπει να σας δώσω τα συγχαρητήρια της Σιλβάνας, όχι μόνο για το έργο αλλά και τη μεγάλη προθυμία που επέδειξε η συγγήτρια καθ' όλη αυτή τη διάρκεια που παρακολουθούμε το θέμα για να στεφθεί με επιτυχία η χτεσινή συνεδρίαση. Επίσης πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά έγιναν διότι η συγγήτρια κατάφερε να φέρει μια απάντηση ισόρροπη που ελάμβανε υπόψη όλα τα θέματα, όλες τις πτυχές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην νομοθεσία γιατί υπάρχουν πολλά συμφέροντα όλα θεμητά και πρέπει να βρεις μια σοφή ισορροπία. Αυτό το έκανε η συγκεκριά. Ε, επίσης έγινε μεγάλος διάλογος και δημοκρατική συνεννόηση μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων ε, η οποία κάθε μια άφησε το στίγμα της εκεί που την ενδιέφερε και είναι πάρα πολύ στεναρή η απόφασή μας τελικά διότι αυτό το θέμα, ξέρετε, είναι πάρα πολύ λεπτό και όλη αυτή η αρχιτεκτονική, η εύθραυστη, ε, ήταν ένα θέμα που μας ενδιαφέρε πάρα πολύ και θέλαμε ε, συγκεκριμένες προθεσμίες για μεταφορά της ε, νομοθεσίας. Ε, έτσι, χωρίς καμία αμφιβολία και με μεγάλο ενθουσιασμό θα υπερψηφίσουμε το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου οι σοσιαλιστές και ελπίζω και την Ολομέλεια περάσει γρήγορα βάσει των νέων κανόνων και άρθρων του κανονισμού έτσι ώστε το 16 να έχει μεταφερθεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Συνεχίστε σε αυτή τη γραμμή, Ελισαμπέτ. Είμαστε μαζί σας. Thank you. Um, the next... Ευχαριστώ. Η Μαριάν Χάρκη. Thank you very much and... Ευχαριστώ πολύ καθώς και την εισηγήτρια για την αποτελεσματική της διαχείριση του θέματος και τον κύριο Θέρκας, όλα αυτά πολύ δημοκρατικά. Η εισηγήτρια προάσπισε τη θέση του Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα ως προς τα μακροπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και τις απαραίτητες εξαιρέσεις που πρέπει να προβλεφθούν, ενώ παράλληλα θέλησε να διασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια όλων των εργαζομένων για την το χρονοδιάγραμμα της μεταφοράς έκανε ό,τι μπορούσε, εργάστηκε σκληρά, καινοτόμησε, συνεννοήθηκε και το μόνο που μπορώ να πω τελικά ως συμπέρασμα είναι ότι είναι εξαιρετική δουλειά. Okay. Um, I give the back the... Καλά, τότε θα ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Λοράνσακη. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ επίσης ειλικρινά τους συναδέλφους που μίλησαν. Ε, ειλικρινά ήταν μια ομάδα εργασίας που λειτουργήσε πολύ καλά γιατί όλοι οι σκιώδεις συνεργάστηκαν ήταν ανοιχτή και έδειξαν μεγάλη θέληση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα Σιλβάνα Ράπτη, τον Γεώργιο Τούσα, Μακιντάι και άλλους. Διότι ποτέ δεν θα καταφέρναμε μια τέτοια δουλειά χωρίς τέτοιο ανοιχτό πνεύμα όλων των σκιωδών. Επίσης πρέπει να πω ότι οι υπηρεσίες της Κομισιόν, η Γραμματεία δηλαδή, μας βοήθησαν πολύ και μας ε, βοήθησαν και οι εμπειρογνώμονες της και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβει κανείς σωστά την προβληματική. Μάλιστα Αλέχανδρε, το κείμενο είναι ισορροπημένο διότι κανείς δεν κατακράτησε πληροφορίες, όλα τα βάλαμε στο τραπέζι και, και αυτό σημαντικό. Εδώ τώρα που τελειώνει αυτή η διαδικασία επί της οδηγίας νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί περήφανοι γιατί ό,τι ζητήσαμε το πετύχαμε για το χρονοδιάγραμμα, για την πληροφόρηση των εργαζομένων, για το σεβασμό της υγείας και ασφάλειάς τους και για τις εξαιρέσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους και όλες και ελπίζω να η ψηφοφορία του απογεύματος να είναι το ίδιο όμορφη. Thank you so much. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως το είπατε θα ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης και θα ψηφιστεί η πρόταση αυτή στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Ας προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης, σημείο 14. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Ντόιτς, είναι εδώ. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την καινοτομία για μια βιώσιμη ανάπτυξη, μια βιοοικονομία για την Ευρώπη. 27 τροπολογίες έχουν υποβληθεί και θα πρέπει να τις εξετάσουμε και δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Ντόιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου δίνετε να συμμετέχω στη συνεδρίαση αυτή με μια κάποια καθυστέρηση, γιατί χρειάστηκε να συμμετάσχω σε μια ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμών. Γι' αυτό το λόγο έφτασα λίγο καθυστερημένος. Όπως είπε η Πρόεδρος, Όντως θα ήθελα να σας μιλήσω εν συντομία για τις 27 τροπολογίες που υποβλήθηκαν στην, στο σχέδιο γνωμοδότησής μου. Η γνωμοδότηση αυτή απευθύνεται στην αρμόδια καθήλυν επιτροπή που είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και η γνωμοδότηση λοιπόν αυτή αναφέρεται στην καινοτομία για μια βιώσιμη ανάπτυξη, μια βιοοικονομία για την Ευρώπη. Το σχέδιο γνωμοδότησης επικεντρώνεται κυρίως στον πολύ σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η βιοοικονομία στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην βιώσιμη επίσης χρήση των πόρων μας, καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση καυσίμων τα οποία δεν είναι ορυκτά καύσιμα. Όπως είπε και η Πρόεδρός μας, έχουν κατατεθεί 27 τροπολογίες από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, από τους Σοσιαλιστές και από τους Φιλελεύθερους. Οι συνάδελφοι οι οποίοι υπέβαλαν τροπολογίες ουσιαστικά δυναμώνουν διάφορες πτυχές της γνωμοδότησής μου και κινούνται στο ίδιο πνεύμα με αυτό που υπάρχει στην Στρατηγική Ευρώπη 2020. Ουσιαστικά τονίζουν ιδιαίτερα το ζήτημα της πράσινης ανάπτυξης και πώς αυτή μπορεί να συμβάλλει σε περισσότερες θέσεις εργασίας και υπογραμμίζουν επίσης τη μετάβαση αυτή από μια οικονομία που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα προς μια οικονομία που θα βασίζεται στην βιοοικονομία. Ουσιαστικά οι τροπολογίε ενισχύουν κάποιε βασικέ ιδέε οι οποίε εκφράζω με την γνωμοδότησή μου. Οι τροπολογίε αυτέ υπογραμμίζουν το ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κυρίως προϊόντα βιολογικής βάσης, ακόμα και από τον τομέα της ξυλίας, και τονίζουν επίσης ότι θα πρέπει η βιοοικονομία να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους νέους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ακόμα πρόοδο προκειμένου να καταφέρουμε να δώσουμε έναν πιο έντονο οικολογικό χαρακτήρα στην βιοοικονομία. Σε καμία περίπτωση θα πρέπει μέσω των δράσεών μας να βάλουμε κατά του περιβάλλοντος. Ένα συνάδελφος επίσης πρότεινε ότι θα ήταν σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να κάνουμε επενδύσεις στην κατάρτιση, στη διαβίου κατάρτιση. Και είπε επίση ότι θα πρέπει να προβλέπεται χρηματοδότηση 25% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την χρησιμοποίηση των ε, πόρων από το Ταμείο Συνοχής. Επίσης προβλέπεται ή προτείνεται μάλλον σε κάθε κράτος μέλος να υπάρχει ένας βαθμός ευελιξίας για τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων αυτών. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας μέσω της βιοοικονομίας και οι θέσεις αυτές εργασίας δεν μπορούν να έρθουν μόνο μέσω των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Είναι Πολύ σημαντικό να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές, οι οποίες θα έρθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα ήθελα να στηρίξω τις ε, τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και θα συνεργαστώ επικοδομητικά με τους συναδέλφους μου, με αυτούς δηλαδή που έχουν υποβάλει τις τροπολογίες αυτές να καταλήξουμε στις συμβαστικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σέρκας. Με ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς, κοιτάξτε, βρισκόμαστε αρκετά κοντά σε όλες αυτές τις ιδέες που μόλις μας παρουσίασε ο Τάμας Ντόιτς. Όπως είπε, οι συνάδελφος Παπαδοπούλου και άλλοι σοσιαλιστές έχουν καταθέσει συνολικά 15 τροπολογίες. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία για να είναι και αυτή η έκθεση ισόρροπη. Η βιοοικονομία κατά την άποψή μας θα πρέπει να θεωρείται ως μια διαδικασία όπου θα λαμβάνεται υπόψη και η εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, ε, των επιχειρήσεων, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι άνθρωποι τους οποίους θίγουν αυτές οι αλλαγές, οι εργαζόμενοι, ε, η κοινωνία. Όταν υπάρχουν αλλαγές πάντα έχεις νικητές ε, και ιτημένους. Θα, πρέπει να προετοιμάζεται αυτή η διαδικασία για να μην ε, υπάρχει ανισομερής κατανομή του κόστους και του ωφέλους αυτής της αλλαγή Γι' αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό που είχε πει ο πρόεδρος Μπαρόσο από το 2001 ε, η ανάπτυξη και η οικολογία θα πρέπει ε, στη βιοοικονομία να συνοδεύονται και από ένα κοινωνικό πυλώνα. Όχι μόνο για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά για να βγάλουμε και ένα καλό αποτέλεσμα από αυτή την οικονομική αλλαγή. Και για μας είναι πολύ σημαντικός ο διάλογος, ο κοινωνικός διάλογος, η διαβούλευση, η κοινωνική εταίρη, οι διαπραγματεύσεις, όλα αυτά να γίνονται με τρόπο συμμετοχικό. Και είναι αυτός ο δρόμος που θα μας οδηγήσει στην επιτυχία και στην ε, εξέβρεση των καλύτερων συνθήκων. Σε αυτή τη βιοοικονομία δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες διαδικασίες που μπορεί να επηρεάζουν ε, την ασφάλεια, την υγεία των εργαζομένων όταν κάπου γίνεται ένα εργοστάσιο πούμε, με, που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματο, αυτό έχει επιπτώσει στου εργαζομένου, στου κατοίκου. Θα πρέπει να τα μελετάμε και αυτά και να τα αντιμετωπίζουμε. Καλή αλλαγή, αλλά θα πρέπει να ε, αξιοποιήσουμε και το ανθρώπινο δυναμικό, γιατί αυτό είναι ο πιο στρατηγικός πόρος στην Ευρώπη που έχουμε εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, διαβίου μάθηση των εργαζομένων, όλα αυτά θα πρέπει να είναι και είναι προς όφελος της κοινωνίας. Ε, τέλος, νομίζω δεν θα έχουμε μεγάλες δυσκολίες να υποστηρίξουμε. Οι δικές μας τροπολογίε φιλοδοξούν η ανάπτυξη αυτή είναι πιο πράσινη, πιο οικολογική και για πρώτη φορά δεν μιλάμε πια στην Ευρώπη για περικοπές και λιτότητα, αλλά πώς μπορούμε να βγούμε προς τα εμπρός νέες ευκαιρίες με αξιοπρεπή ζωή και σεβασμό ε, του κοινωνικού πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ε, όραμα της κοινωνικής οικονομίας αγοράς που χαρακτηρίζει την Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χάρκιν. Thank you. Uh, my colleague... Ευχαριστώ. Πρέπει πάλι να αντικαταστήσω τον συνάδελφο που μου ζήτησε να διαβάσω τις παρατηρήσεις του. Πρώτον ευχαριστή για την εισήγηση και τους υπόλοιπους συναδέλφους για τις τροπολογίες τους. Συμφωνεί με πολλές από αυτές. Είναι φανερό ότι όλοι οι συνάδελφοι αναγνωρίζουν τη σημασία του τομέα η τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Συμφωνεί με το πρώτο τμήμα για την ανάγκη αναπτύξης δεξιοτήτων ιδιαίτερα επαγγελματικής κατάρτισης και μετεκπαίδευσης, ε, ιδίως στην Ήπεθρο. Παρόλα αυτά, οι τροπολογίες στην ε, έκθεση Δίας Πρωτοβουλίας Θέρκας δεν έχουν σχέση με την κεντρική ιδέα της ε, γνωμοδότησης. Επίσης, για την τροπολογία 15 της κυρίας Παπαδοπούλου θα ήθελε να ρωτήσει Υπάρχουν αμφιβολίες προς το πόσες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020 και ευχαριστεί εκ νέου για την εισήγηση και αναμένει τα επικοδομητικά σας σχόλια. Ευχαριστούμε. Τώρα η Κομισιόν, ο κύριος Ντούντ. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει το ενδιαφέρον που δείχνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στρατηγική βιοοικονομίας και για την υποστήριξη που μας δείχνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στρατηγική μας αυτή. Και χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την εμπλοκή τη δική σας επιτροπής καθότι η κοινωνική διάσταση είναι πολύ σημαντική για την στρατηγική βιοοικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό τονίζεται τόσο στο σχέδιο γνωμοδότησης όσο και στις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με το όραμα της δικής σας Επιτροπής ότι η βιοοικονομία μπορεί και θα πρέπει να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ότι θα πρέπει να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη των, της υπαίθρου, των παράκτων περιοχών και συμφωνούμε ότι οι επενδύσεις στις νέες δεξιότητες, στην ανάπτυξη των νέων δεξιότητων σε διάφορα επίπεδα είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να καταφέρουμε να ενισχύσουμε το δυναμικό της βιοοικονομίας. Εκτιμούμε κάποιες από τις ιδέες και τις νέες ιδέες που έχουν υποβληθεί μέσω τροπολογιών. Δεν, έχουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα σχόλια. Ως προς το τελευταίο αυτό θέμα, όσον αφορά δηλαδή την δημιουργία θέσεων εργασίας από το Horizon 2020, θα μπορούσαμε στο μέλλον να δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες γραπτό στη γραμματεία της Επιτροπής, αν επιθυμείτε κάτι τέτοιο. Thank you for Ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα πάλι έχει ο κύριος Ντόιτς, ο συγητής μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι, που υποβάλατε όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσε ιδέες. Θα επαναλάβω κάποια πράγματα τα οποία ακούσαμε και σήμερα το πρωί. Όλοι όσοι πήραν το λόγο έχουν υποβάλει τροπολογίες. Όλοι όμως συμφωνούν με τις βασικές ιδέες της ε, γνωμοδότησής μου. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Δεν θα ήθελα λοιπόν να επαναλάβω όλες αυτές τις προτάσεις. Ωστόσο, θα λάβω υπόψη τις προτάσεις σας προκειμένου να αντικατοπτρίζονται τελικά στο τελικό σχέδιο της γνωμοδότησης και αυτό θα βοηθήσει τελικά στην γενικότερη έγκριση της ε, γνωμοδότησης αυτής και θα συμβάλλει στην στρατηγική βιοοικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντόιτς. Θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότησή σας στην Επιτροπή μας στις 7 ε, Μαΐου Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 19 της ημερήσιας διάταξης. Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Δίνω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Μογάν Σαχτιέ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι πολύ πιο χρονοβόρες και δύσκολες από ό,τι για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ευτυχώς που τουλάχιστον ένας τριμερής διάλογος βαίνει γιατί για τον συγκεκριμένο αυτό τριμερή διάλογο στο οποίο θα σας μιλήσω θα πρέπει να δείξουμε αρκετό κουράγιο και δύναμη. Χθες το βράδυ είχαμε την 15η κατά σειρά συνεδρίαση στα πλαίσια τριμερούς διαλόγου και μάλιστα συνεδράσαμε μέχρι αργά το βράδυ. Πρέπει να σας πω επίση ότι την προηγούμενη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια τη 14 η συνεδρίασής μας, μάλλον ε, ο 14ος τριμερής διάλογος διεκόπη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αποχώρησε τελικά, γιατί δεν συμφωνούσε καθόλου με τον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετώπιζε το Συμβούλιο, το οποίο δεν εκτιμά καθόλου ούτε σέβεται το ρόλο του συνομοθέτη που έχουμε. Από ό,τι φαίνεται, το Συμβούλιο δεν θέλει να αποδεχθεί ότι από την συνθήκη τη Λισαβόνα και μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλέον έχει αυξήσει αρμοδιότητέ του και είναι συνομοθέτη σε πολλού νέου τομεί. Στον 14ο τριμερή λοιπόν διάλογο, το Συμβούλιο έθεσε ένα αμφιβόλο εκ νέου όλε τι συζητήσει που είχαμε κάνει στο παρελθόν κατά τη διάρκεια τη Κυπριακή Προεδρία. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορούσαμε να το αποδεχτούμε σε καμία περίπτωση. Άρα, ζητήσαμε να γίνει ένα τρεμερής διάλογος υψηλού επίπεδου πλέον, για να καταφέρουμε να συζητήσουμε με άλλους ανθρώπους και όχι με την ομάδα διαπραγμάτευσης του Συμβουλίου, αυτή που προβλέπεται αυτή τη στιγμή, γιατί η ομάδα αυτή όχι μόνο δεν σέβεται το καθεστώς της συναπόφασης, αλλά η όλη διαπραγμάτευση είναι μη συμμετρική με το Συμβούλιο. Δηλαδή εμείς, η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από όλε τι πολιτικέ ομάδε και χάρη στην ψηφοφορία τη Επιτροπή μα Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική εντολή για τη διαπραγμάτευση. Και απέναντί μα έχουμε διοικητικού ουσιαστικά υπαλλήλου Συμβουλίου που δεν έχουν καμία απολύτω πολιτική εντολή και που περιμένουν τελικά να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει για το σύνολο του κειμένου, προκειμένου να επιστρέψουν στα κράτη-μέλη και να τα ενημερώσουν. Εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Συνεπώς, η Πρόεδρός μας, η Περβόνς Μπερές, και πρέπει να σας πω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν για όλα αυτά τα σημεία. Ε, υπάρχει πολύ μεγάλη λεγγύη ανάμεσά μας. Η Περβόνς Μπερές, λοιπόν, μετά την διακοπή των διαπραγματεύσεων, ήρθε σε επαφή τηλεφωνικά με τον πρέσβη Μονγκόμερη και του ζήτησε να διεξαχθεί ένα τριμερής διάλογος υψηλού επίπεδου, όπου θα έχουμε την ομάδα διαπραγμάτευσης απασχόλησης και από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους πρέσβεις και το άλλο προσωπικό το οποίο προβλέπεται από το Συμβούλιο. Γιατί όπως σας είπα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με το εφιστάμενο σχήμα. Καταφέραμε μία κάποια πρόοδο να την πετύχουμε, αλλά ουσιαστική διαπραγμάτευση δεν έχει γίνει. Όσον αφορά το άρθρο 3, δεν κάναμε τίποτα παραπάνω από ό,τι προβλεπόταν τελικά, γιατί δεν έχουμε καταλήξει αυτή τη στιγμή σε καμία γενική συμφωνία. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία επίσης για το άρθρο 4. Και το άρθρο 4 είναι πραγματικά η ουσία του ζητήματος. Ασχολούμεθα στο άρθρο 4 με τα πιο ευαίσθητα ζητήματα, αυτά δηλαδή αυτά τα που μας απασχολούν περισσότερο. Δηλαδή, τι θα γίνει με το 25% της χρηματοδότησης προβλέπεται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ζητήσαμε επίσης να υπάρχει ένας οδικός χάρτης για τη διαπραγματευτική ομάδα, αλλά και πάλι μας δώσαν απλώς κάποια στοιχεία και κάποια δεδομένα, τίποτα το τόσο ουσιαστικό. Και χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, επιμείναμε στις τροπολογίες εκείνες οι οποίες είναι ακόμα προβληματικές, αυτές που εκκρεμούν. Και συνοψίζοντας, πρέπει να σας πω τα ακόλουθα, ότι έχουμε πέντε σημεία, τα οποία είναι ιδιαίτερα λεπτά και ευαίσθητα. Το πρώτο έχει να κάνει με τον τίτλο Εμείς στηρίζουμε τον τίτλο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι αυτόν που προτείνει το Συμβούλιο. Δεύτερο σημείο. Τροπολογία 40. Όσον αφορά την βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση που ανταποκρίνεται στις γραμμές προσανατολισμού για την στρατηγική 2020, τροπολογία 54 όσον αφορά την ενεργή ένταξη τροπολογία 59 όσον αφορά τα δύο φύλλα και την τροπολογία 61 όσον αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, όπου για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το Συμβούλιο μας έλεγε δίθεν ότι δεν γνώριζε καν τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Και χθε το βράδυ πραγματικά με σόκαρε Κοιτάξτε, πώς να σας το πω. Σχεδόν ψέματα μας λέγανε οι άνθρωποι του Συμβουλίου. Αυτοί δηλαδή που συμμετέχουν στη διαπραγματευτική ομάδα του Συμβουλίου. Δηλαδή, ενώ υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, τα παρουσίαζαν όπως τους βόλευαν. Χειραγωγούσαν κάποια στοιχεία δηλαδή για να τα παρουσιάσουν προς όφελός τους. Απόλυτα ψεύδι λοιπόν όπως καταλαβαίνετε. Ω εκ τούτου, η διαπραγμάτευση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους και συγητές, οι οποίοι δείξανε μια πολύ επικοδομητική στάση και όλους ιδιαίτερως να ευχαριστήσω την Κίνκα που είναι εδώ μαζί μας και η οποία πρότεινε μια νέα διατύπωση για τον τίτλο όσον αφορά την ενεργή ένταξη ενσωμάτωση γιατί από τη μια εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε την ενεργή ενσωμάτωση όλων των ανθρώπων, ο τίτλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άλλωστε είναι «Ενεργή ένταξη, ενεργή ενσωμάτωση», ενώ το Συμβούλιο πρότεινε την ενεργή ένταξη με ιδιαίτερο στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας. Και τι κρυβόταν πίσω από αυτό. Το Συμβούλιο ουσιαστικά, τα κράτη-μέλη δεν ήθελε την ενεργή ένταξη όλων των πολιτών ήθελε ουσιαστικά να επικεντρωθεί η ενεργή συμμετοχή προς τους ε, άνεργους για να επιστρέψουν αυτοί σε καθεστώς απασχόλησης. Ουσιαστικά τα κράτη-μέλη θέλουν να χρησιμοποιήσουν ε, την περίφημη ενεργή ενσωμάτωση μόνο και μόνο για να μειώσουν τα ποσοστά ενεργείας που έχουν στις χώρες τους. Χάρη λοιπόν σε μια νέα διατύπωση, την οποία μπορώ να σας διαβάσω και αργότερα αν θέλετε, καταφέραμε να ξεπεράσουμε το προβληματικό αυτό σημείο και τελικά καταφέραμε να σημειώσουμε πρόοδο και στα υπόλοιπα σημεία. Αυτά είχα να σας πω κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Η Κίνγκα. Ευχαριστώ πολύ. Η Ελισάβετ μας τα είπε πολύ καλά. Η διαδικασία βέβαια είναι αρχή και μακρόσυρτη. καθόμασταν μέχρι και τα μεσάνυχτα γιατί θέλαμε να καταλήξουμε κάπου. Το κύριο θέμα και ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα καταμοιραστεί, θα κατανεμηθεί το ESF, το Κοινωνικό Ταμείο τα κονδύλια του. Εμείς είμαστε πεπισμένες ότι μόνον αν καθοριστούει η κατανομή αυτή μόνο τότε θα πιστούν τα κράτη-μέλη γιατί έχουν φοβερές αντιστάσεις. Σε συναντήσεις υψηλού επίπεδου υπουργικού, στο Συμβούλιο δηλαδή με επιτρόπους, φαίνεται ότι And it also the ESF share is... φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό πρόβλημά τους το CPR που λένε. Προσπαθήσαμε λοιπόν να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία και γι' αυτό σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Ταυτόχρονα επεξεργαζόμαστε τις λεπτομέρειες και τους στόχους. Εχθές κάτι καταφέραμε, αλλά δεν είναι εύκολο να συνεργάζεται κανείς με το Συμβούλιο. Και στην Επιτροπή ΕΛΕΦ προσπαθήσαμε να ζητήσουμε συνεννόηση αλλά δεν είναι όλοι οι τριμερείς διάλογοι τόσο δύσκολοι όπως αυτός γι' αυτό είμαστε αισιόδοξοι ότι μετά την συνάντηση ψηλού επίπεδου θα διευκολυνθούν τα πράγματα. Α, μάλιστα. Θέλετε να ξαναμιλήσετε. Κοιτάξτε, το 25% των ταμείων συνοχής που θα κρατηθούν στο κοινωνικό ταμείο για μας είναι θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει, το αγώνα θα είναι δύσκολος. Πρέπει να σεβαστούμε απολύτως αυτό το μερίδιο των ταμείων συνοχής με βάση τα κοινωνικά θέματα. Αλλιώς η κοινωνική Ευρώπη θα αμφισβητηθεί από τα κράτη-μέλη. Και στη διαπραγματευτική μας ομάδα ούτε ένας σκιώδης δεν θα παρετηθεί από αυτό το αίτημα. Ούτε ένας. Α, ναι, ναι σωστά. Σας κατευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα το επόμενο θέμα, το 20, διαπραγματεύσει με το συμβουλή σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, έτυπε. Η εισηγήτριά μας Μάριν Χάκιν, σαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομη θα είναι η συζήτηση γιατί Κάναμε έναν πρώτο τριμερή διάλογο στο Στρασβούργο με το Συμβούλιο και την Κομισιόν, αλλά δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε, διότι η μπλοκαριστική μειοψηφία στο Συμβούλιο υπάρχει ακόμα και δεν υπήρξε συμφωνία λοιπόν. Η επόμενη συνάντηση του Κορεπέρ είναι 2 Μαΐου περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει, αν θα σημειωθεί καμία πρόοδος εκεί. Είναι πολύ απογοητευτικά όλα αυτά βέβαια γιατί είχαμε συμφωνήσει προηγουμένως αλλά δεν έγινε καμία πρόοδος επί των συμπεφωνημένων. Τα τρία θέματα που παραμένουν όπου δεν υπάρχει συμφωνία λοιπόν είναι το κριτήριο για την κρίση, το εύρος του κανονισμού, δεύτερον η ρυθμίση χρηματοδότησης και τρίτον ο ορισμός του εργαζομένου. Όλα αυτά είναι απογοητευτικά διότι δεν ε, έγινε καμία ουσιαστική πρόοδος και για τα τρία αυτά. Έγινε μια άτυπη συζήτηση μετά τη συνάντησή μας με την Κομισιόν και εκείνοι ανησυχούν γιατί δεν σημειώθηκε πρόοδος και συμμερίζονται τις, ίδιες, τις δικές μας ανησυχίες. Δεν μπορώ να σας πω τίποτε άλλο, πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 2 Μαΐου. Θα ήθελα να ακούσω αν οι συνάδελφοι έχουν καμιά ιδέα, αλλά μέχρι τώρα περιμένουμε. Και δεν ξέρουμε ούτε καν τι περιμένουμε. Α, ωραία. Μήπως θέλει κανείς να μιλήσει. Όχι. Καλά. Ευχαριστούμε Μάριον για όσα μας έχεις κάνει. Πάμε τότε στο επόμενο θέμα. Ποιο είναι το επόμενο θέμα. Δεν έχει τελειώσαμε. Ω, ωραία. Ε, τότε θα ξανασυναντηθούμε το απόγευμα.